Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι στη διάθεσή σας. Εάν υπάρχουν σχόλια, αλλά δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω, επομένως εγκρίνονται τα πρακτικά. Και σας ευχαριστώ. Έχουμε δύο θέματα να, συνεχίσουμε, να συζητήσουμε σήμερα επί του προϋπολογισμού. Το πρώτο